78 του κανονισμού την ευκαιρία να υπογράψουμε μια, ένα κοινό κείμενο για την τακτική νομοθετική διαδικασία με κείμενο το οποίο θα προσαρτηθεί στα πρακτικά της